Κυρίες και κύριοι, άρχεται συνεδρίασης. Πρώτο σημείο της ημέρας της διάταξης, η έκθεση Μπαλτσάνη. τριμερής διάλογος, η εντολή μάλλον επί του τριμερούς, διαλόγου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2004. Έχει το λόγο για 4 λεπτά η συγκίτρια κυρία